Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε, ήφιστε να περιμένουμε την ολοκλήρωση της διάσκεψης των Προέδρων πρώτου ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Προκαταρκτικά να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Ροζάριο Κροτσέτα, πρώην βουλευτής του Κοινοβουλίου, απίφθινε στον Πρόεδρο αίτηση για την προάσπιση της βουλευτικής του ασυλίας στα πλαίσια μιας προδικαστικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Παλέρμο. Βάση του κανονισμού αποστέλλεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου το θέμα, η οποία είναι και καθήλυνα αρμόδια.